Καλημέρα. Καλά δεν είναι και τρομακτική προσέλευση. Ε, ξέρω ότι δυσκολεύεται ο κόσμος να βρει την αίθουσα και να συρθεί μέχρι εδώ. Αλλά ας αρχίσουμε σιγά σιγά. Είναι κοινή συζήτηση για την ε, οδηγία για την πρόληψη τη χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικού συστήματο για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Και είναι επίμαχο αν εμεί είμαστε αρμόδιοι επί τη ουσία ή όχι επιτροπή. Γιατί πρόκειται για την τροποποίηση της οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματο, και αυτό είναι μάλλον οικονομικά ζητήματα και λιγότερο ελευθεριών είναι νομικό. <laughs> Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν έχει λυθεί. Συνεχίζεται αντιπαράθεση. Θα δώσω το λόγο στους ε, συντάκτες νομοδότηση στου συζητητέ ανάλογα. Ποιος ε, θα τύχει, ο κύριος Κάριν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στην χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματο για νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε και χρηματοδότηση τρομοκρατία. Επομένω, στο λογικό θα ήταν εμεί να ήμασταν η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Θα δούμε όμω πώ εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Υπολογίζεται ότι η νομοποίηση εισόδων από παράνομε δραστηριότητε αντιστοιχεί περίπου στο 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. και θα έλεγα ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν υπέβαλε μία πρόταση προκειμένου ο κανονισμός να γίνει πιο αυστηρός, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της νομοποίηση εσόδων παράνομων δραστηριότητε και να περιοριστεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατία και των ε, παράνομων ε, δραστηριοτήτων. Ένα μέτρο προβλέπεται ω προ αυτό είναι το μέτρο το οποίο ονομάζεται beneficial ownership, δηλαδή ποιο είναι ο τελικός ουσιαστικός δικαιούχος των χρημάτων που έχουμε σε ένα λογαριασμό ή σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, οι εμπλεκόμενοι, για παράδειγμα ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και το καθεξής, είναι οι υπεύθυνοι. Αυτοί πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι ο πελάτης τους. Έτσι λοιπόν λειτουργούσαν τα πράγματα μέχρι σήμερα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τώρα να προβλέπονται και κάποιοι νέοι τομεί, όπω για παράδειγμα το μέσο των τυχερών παιχνιδιών, ο οποίο παρουσιάζει αύξηση ιδίω στα πλαίσια του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, στο διαδίκτυο και που θεωρείται ένα τομέα στον οποίο λοχεύουν κίνδυνοι όσον αφορά την νομοποίηση εισόδων παράνομε δραστηριότητε επίσης καλύτερη παρακολούθηση, μείωση από 15.000 σε 7.000 των χρημάτων που μπορούν ηλεκτρονικά να μεταφερθούν με εμβάσματα, νομίζω ότι όλα αυτά τα μέτρα κινούνται προς σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ωστόσο ότι το να είναι μεμονωμένες εταιρείε, επιχειρήσεις ή οντότητες υπεύθυνε για το ποιος είναι τελικός δικαιούχος είναι κάπως προβληματικό. Θεωρώ ότι κάθε κράτος μέλος έχει ένα μητρό επιχειρήσεων. Προκειμένου να δραστηριοποιηθεί κανείς επιχειρηματικά θα πρέπει να καταχωρήσει σε ένα εθνικό μητρό την επιχείρησή του και αν καταφέρουμε εμείς να βελτιώσουμε τη φυστάμενα αυτά εθνικά μητρώα, αν καταφέρουμε δηλαδή να έχουμε στα πλαίσια των εθνικών μητρώων τους τελικούς δικαιούχους μιας επιχείρησης, τότε θα σημειώναμε ένα τεράστιο βήμα πρόοδου, χωρίς να χρειάζεται ουσιαστικά να τροποποιήσουμε το φυστάμενο σύστημα. Έχουμε ήδη μια οδηγία, την 70 του 2012, 17 με συγχωρείτε, του 2012, που αναφέρεται στην ε, δυνατότητα σύνδεσης αυτών των εθνικών μητρώων. Θεωρητικά θα έπρεπε σύμφωνα με την οδηγία αυτή να είναι στεδεμένα τα μητρώα αυτά, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει ακόμα στην πράξη. Θα μπορούσαμε λοιπόν να λέμε ότι στα πλαίσια των ίδιων των μητρών θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι ο τελικό δικαιούχο, προκειμένου να μπορεί μια επιχείρηση να λειτουργεί. Αν καταφέρναμε να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο, νομίζω θα μειώναμε σε σημαντικό βαθμό τις παράνομες αυτές συναλλαγές και θα μπορούσαμε επίσης να γνωρίσουμε με ποιους συνδιαλέγονται και με ποιους συνεργάζονται οι επιχειρήσεις. Στη συνέχεια υπάρχει ένα άλλο θέμα. Πρέπει να είναι δημόσια τα μητρώα αυτά ή θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο οι αρχές κάθε χώρας. Νομίζω ότι όσον αφορά τις ε, διοκτικές αρχές και τις ε, φορολογικές αρχές μιας χώρας, αυτές προφανώς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα μητρώα αυτά. Αν τα μητρώα βέβαια αυτά ήταν εντελώ δημοσίω ανοιχτά, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά και για του ίδιου του ε, εγκληματίε, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιλέξουν στη συνέχεια σε ποια επιχείρηση θα απευθυνθούν ή θα μπορούσαν τουλάχιστον να παρακάμψουν τα μέτρα τα οποία προβλέπονται σε ένα κράτος μέλος. Νομίζω λοιπόν ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εισάγουμε το νέο αυτό σημείο, το οποίο βελτιώνει και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον τώρα, Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τα όσα λέγονται για την αξιολόγηση του κινδύνου, την εκτίμηση του κινδύνου. Και αυτό όσον αφορά την κατανομή των κεφαλαίων. Καταλαβαίνετε ότι ε, η κατανομή των κεφαλαίων θα πρέπει να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, οι ε, πόροι αυτοί βάσει εκτίμηση κινδύνου για την καταπολέμηση τη νομοποίηση εισόδων από παράνομε δραστηριότητε. Πρέπει δηλαδή εξ αρχή να δούμε ποιε δραστηριότητε ελοχεύουν περισσότερου κινδύνου και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι απαραίτητοι πόροι προκειμένου να περιοριστούν οι δραστηριότητε αυτέ βάσει εκτίμηση κινδύνου. Νομίζω θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την ιδέα αυτή. Και τέλος, θα ήθελα να αφαιρθώ στο ζήτημα του ανταγωνισμού. Από προσωπική πείρα πριν από μερικά χρόνια ίδρυσα μια εταιρεία στην Λετωνία που από την παραγωγή πάγους προχώρησε στο να γίνει τελικά μια εταιρεία κατεψυγμένων προϊόντων. Είδαμε ότι, είδα στη δική μου την περίπτωση ότι πολλές φορές ο ανταγωνισμός ήταν τόσο πιεστικός που χρειάστηκε για κάποια προϊόντα να κατεβώ και κάτω από την τιμή του κόστους και κάποιες εταιρείες προχωρούσαν σε πολύ χαμηλότερη τιμή και δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μπορούσαν να χαμηλώνουν τόσο πολύ τις τιμές των προϊόντων τους. Τη στιγμή που καταβάλαμε τους ίδιους μισθούς το ίδιο ποσοστό φορολογίας, πληρώνουμε το, το ίδιο ποσό όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα για παράδειγμα. Και έμαθα λοιπόν πριν από μερικά χρόνια όταν κάποιος ανταγωνιστής μου αποφάσισε να πουλήσει την εταιρεία του, ότι ε, ο ανταγωνιστής τελικά αυτός μου δείξε τα πραγματικά του περιουσιακά στοιχεία. Ουσιαστικά είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια επιχείρηση η οποία δεν κατέβαλε φόρους και κατά αυτόν τον τρόπο κατάφερνε να μειώσει πάρα πολύ τις τιμές του ακριβώς επειδή το κόστος, το κόστος του ήταν 20% χαμηλότερο από το δικό μου. Πώς θα μπορούσα εγώ ποτέ να ανταγωνιστώ κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα με την φοροδιαφυγή και την νομοποίηση εισόδημα παράνομες δραστηριότητες είναι ότι πολλές φορές τα φαινόμενα αυτά βασίζονται σε τέτοιες άτυπες παράνομες οικονομικές δραστηριότητες που επηρεάζουν πάρα πολύ και τις ίδιες επενδύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε λοιπόν πώ ε, γίνονται οι επενδύσεις αυτές και τελικά υπάρχει ένα ισότιμο ανταγωνιστικό πεδίο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιε επιχειρήσει οι οποίε μπορούν να παρακάμπτουν το φορολογικό σύστημα και υπάρχουν άλλε επιχειρήσει παράλληλα οι οποίε είναι μικρομεσαίε και οι οποίε δεν έχουν του απαραίτητου πόρους προκειμένου να αποφύγουν τη φορολογία, τότε καταλήγουμε στο να έχουμε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες εντελώς παράνομα προωθούνται, ε, βρίσκονται σε προνομιούχα θέση και ξέρετε ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ ακόμα και τη δημιουργία των θέσεων εργασία, γιατί ξέρετε ότι είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αυτέ οι οποίε προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό θέσεων απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι σιγά σιγά, τουλάχιστον στη δικιά μου τη χώρα, οι επιχειρήσει αυτέ οι οποίε καταφέρουν να μην καταβάλουν φορολογία εξαφανίζονται σιγά σιγά. Αν δούμε όμω πιο σφαιρικά το ζήτημα αυτό, βλέπουμε ότι η οδηγία αυτή προσπαθεί να αντιμετωπίσει και αυτό το φαινόμενο. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για την αντιμετώπιση τη νομιμοποίηση εσόδων παράνομε δραστηριότητε, αλλά και για την ίδια την φορολογία των επιχειρήσεων να δημιουργηθεί ένα καλύτερο επίπεδο ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να καταφέρουμε να προσελκύσουμε και περισσότερε επενδύσει. Αν, αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλο και περισσότερε επιχειρήσει θα καταβάλουν εφόρου και ότι θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τελικά ποιο είναι ο δικαιούχο των επιχειρήσεων κάθε φορά που γίνονται πληρωμέ, για παράδειγμα, θα βελτιώσουμε πάρα πολύ τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να φερθώ σε αυτά τα ζητήματα στη δική μου τη γνωμοδότηση. Α καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε στα πλαίσια των εθνικών μετρών ποιο είναι ο δικαιούχο, αυτό το οποίο στα αγγλικά ονομάζουμε beneficial ownership. Και επίση πρέπει να σα πω ότι υποστηρίζω ιδιαίτερα την προσέγγιση με εκτίμηση κινδύνου που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για λόγου ισότιμου ανταγωνισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια τη οδηγία αυτή να καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη συμμόρφωση με την καταβολή φόρων, για την καταβολή φόρων, με συγχωρείτε, και μέσω κάποιων νομοθετικών τροποποιήσεων νομίζω ότι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε το κλίμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως σας είπα είναι αυτές που δημιουργούν τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κλέβα που είναι συντάκτη γνωμοδότης της δεύτερης έκθεσης. Ευχαριστώ πρόεδρε, δεν κατάλαβα ότι ήταν κοινή η συζήτηση. Λοιπόν, συμπληρωματικό με το ξέπλυμα χρημάτων και τη τρομοκρατία έχουμε ε, τώρα πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και τον αντίστοιχο κανονισμό. Ε, τι στόχο έχει ο νέος κανονισμός να ε, βελτιωθεί η διαφάνεια στα εμβάσματα κάθε είδους, εγχώρια και διασυνοριακά, για να μπορούν οι διοκτικές αρχές ε, να εντοπίζουν περιπτώσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος και τρομοκρατίας. Ο σαφέστερος σύνδεσμος μεταξύ των δύο θεμάτων ποιος είναι είναι οι βασικές προφορίες για ε, εκείνον που ε, κάνει τη μεταφορά ε, των χρημάτων, εκείνος που δίνει την εντολή δηλαδή για το έμβασμα, να μπορεί άμεσα να εντοπίζεται από τις διοκτικές αρχές, για να εντοπίζονται και όλες του οι Είναι κανονισμός αντίστοιχος με την οδηγία και προσαρμόζεται στα διεθνή πρότυπα. Οι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν ε, προσπαθούν να βελτιώσουν ε, την ε, ειχνηλασιμότητα των πληρωμών. Βέβαια, διαβεβαιώνοντας ότι το πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα διεθνώς ισχύοντα για την, από την ομάδα δράσης που δημιουργήθηκε πέρσι για την χρηματοπιστωτική δράση. Βασικά είναι ο μεγάλος αδελφός, ο μικρός αδελφός τεχνικός, ο μικρός αδελφός του μεγάλου. Λοιπόν, είναι ένα καλό σήμα, ε, είναι καλό μήνυμα, ε, δεν έχουμε μεγάλες δυσκολίες στην εφαρμογή. Από την άλλη όμως, ε, θα ήθελα να πω ότι Παρόλο που ο κανονισμός μένει σε αρκετά τεχνικό επίπεδο, θα πρέπει να υπάρχει και να εξασφαλίσει συνέπεια και συνέχεια μεταξύ των δύο συναφών αυτών θεμάτων. Να μην έχουμε κανένα διαβολάκο εκεί να κρύβεται στις λεπτομέρειες του κανονισμού. Σε σχέση με την αρχική συζήτηση που γίνεται σήμερα, θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά ζητήματα. Τα είπε μερικά ο κύριος Κάνης, αλλά είναι πιο τεχνικά δικά μου. Ε, η ΦΑΤΑΦ, δηλαδή η ομάδα δράσης αυτή, κάνει μια επισκόπηση των διεθνών προδιαγραφών και καλό είναι για να παρακολουθούμε και τις αλλαγές στο ξέπλυμα ε, και τη χρηματοδότηση. Οι τάσεις αλλάζουν και τα τεχνολογικά μέσα ε, που έχουν στη διάθεσή τους οι εγκληματίες για τις εγκληματικές δραστηριότητες. Οι νέες λοιπόν προδιαγραφές είναι κάτι που παρακολουθούμε έτσι ώστε, ε, σας είπα, το δικό μας νέο πλαίσιο να συνάδει με το αναφερειμένο διεθνές. Να παρακολουθεί λοιπόν και το ευρωπαϊκό πλαίσιο της εξελίξης, γιατί πραγματικά δεν έχει όρια η εφευρετικότητα των κακοποιών σε αυτά τα συστήματα και θα πρέπει ε, από παντού εμείς να ε, φροντίσουμε να τα κλειδώνουμε ώστε να μην υπάρχουν παραθυράκια ο δικός μου είναι κανονισμός, η άλλη λοιπόν είναι οδηγία και για τα εμβάσματα και τις μεταφορές χρηματικών ποσών θα πρέπει να έχουμε πληροφορίες και για εκείνον που στέλνει τα χρήματα και για εκείνον που τα παραμβάνει, που είναι τελικός αποδέκτης. Και οι ε, διοκτικές αρχές και οι άλλες αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν κάθε ε, πληροφόρηση για να μπορούν αποτελεσματικά να καταπολεμούν την ε, νομιμοποίηση εισόδων από παράνομους δραστηριότητες. Ε, υπό το φως λοιπόν και της ενιαίας αγοράς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ζητεί πληροφορίες μόνο για εκείνον που δίνει την εντολή ε, και όχι για εκείνον που λαμβάνει το ποσό. Αλλά επειδή έχουμε εδώ θέματα φοροδιαφυγής και φοροαπαλλαγής, άρχισα να αναρωτιέμαι για την καταπολέμηση και του ξεπλήματος εκτός από τη φοροδιαφυγή, μήπως θα μπορούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ασχολούμαστε όχι μόνο με εκείνον που εμβάζει τα χρήματα, αλλά και με εκείνον που τα παραλαμβάνει. Ε, είναι γεγονό ότι ε, αυτό είναι σημαντικό και θα ήθελα να ακούσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γνώμη έχει. Το επιχείρημα της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό, αλλά να κοιτάμε τι γίνεται και με τους δικαιούχους, με τους αποδέκτες, για να είμαστε αποτελεσματικοί στην ε, καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος, του ξεπλήματος και της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο, το είπε και ο προηγούμενος ε, εισηγητής. Ανησυχώ λίγο σε σχέση με τον ορισμό της ασάφειας σε σχέση με την προσέγγιση με βάση τους νέους κινδύνους. Δηλαδή, τι εννοώ. Είναι διαφορετικός ο κίνδυνος για τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Άρα, μια πιο υπεύθυνη προσέγγιση θα έχει και καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο μεγάλες τράπεζες ε, που θα κάνουν σωστή ανάλυση κινδύνου, αλλά θα πρέπει και τα μικρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μη χρηματοπιστωτικά, ας πούμε, δικηγορικές εταιρείες, οι δικηγόροι να καλύπτονται από αυτό, για να υπάρχει μια καλή ισορροπία, να υπάρχει σωστή ανάλυση του κινδύνου και σωστή αντιμετώπιση από όλους τους φορείς και να είναι αυστηροί οι κανόνες για να ισχύουν προς πάσα κατεύθυνση. Επίσης, ανησυχώ ε, για τις κυρώσεις ε, τι γίνεται με τα μικρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί υπάρχει μια νομική ασάφεια, ένα θολό τοπίο ε, και αφήνεται ανοιχτό ε, στη σημερινή εκδοχή του κανονισμού και χωράει βελτίωση πολύ. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω ε, στην έκθεσή μου είναι ε, ο κανονισμός ΣΕΠΑ, ε, η οδηγία για τις πληρωμές και για τη μεταφορά πιστώσεων, ποιες είναι οι διαφορές αυτά τα νομοθετήματα και θα ήθελα τα δικά σας σχόλια και ενδεχομένω και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Indeed, Mrs. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κλέβα ο εξ των ε, σοσιαλιστών. Ο κύριος Σίμων, ευχαριστώ. και τους δύο συγκητές, πάρα πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπαν. Συμφωνούμε όλοι για την καταπολέμηση του ξεπλήματος και την καταπολέμηση των ε, φορολογικών ε, εγκλημάτων θα πρέπει να τους κοπεί ε, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και για την τρομοκρατία. Ε, αλλά υπάρχουν και άλλοι, δεν είναι μόνο οι τράπεζες, ε, είναι και το καζίνο και οι δικηγόροι, όλοι αυτοί δεν ξεπλένουν χρήματα για εγκληματίες, τους χρειαζόμαστε. είναι φορείς με τους οποίους πρέπει να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε το θέμα της καταπολέμησης του ξεπλήματος. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουμε πάντα ποιος είναι ο συνομιλητής, η ταυτότητά του. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος είναι ο τελικός οικονομικός δικαιούχος πίσω από μια ε, εμπορική συναλλαγή. Ε, για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά χρειάζεται πολύ καλή πληροφόρηση με στοιχεία που θα πρέπει να συλλέγουν αλλά και να τηρούν. Ε, και θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται, αλλά δεν σημαίνουν τεράστια επιβάρυνση όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά κυρίως για ε, ανθρώπους που υποχρεούνται να το πράττουν χωρίς να είναι οικονομικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δηλαδή, να μην εμποδίζουν τη λειτουργία τους αυτές οι απαιτήσει που τους θέτουμε. Και επίση τι κάνουμε με τα δεδομένα και τα οικονομικά στοιχεία από τρίτες χώρες. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι ε, η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο ε, μπορεί να αντιμετωπίσει το ξέπλυμα ιδιαίτερα σε ευαίσθητες συναλλαγές, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τους εξής δύο λόγους και με κανόνες και με οδηγίες. Ε, να μην έχουμε ε, αυθαιρεσίες ή διάφορες εφευρέσεις θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμόνιση αν θέλετε ή μια ε, κάποια στοιχειώδη δυνατότητα συντονισμού των συστημάτων. Για να μην μπορεί ο κακοποιός να ε, επιλέγει από 27 διαφορετικά συστήματα εκείνο που το ε, συμφέρει περισσότερο. Και επίση αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μην επιβαρύνουμε ιδιαίτερα ε, τους φορείς και οι ελάχιστε προδιαγραφές προς τα κάτω να ε, είναι σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Ένα τελευταίο για τον τζόγο, τα τυχερά παιχνίδια. Καταρχήν, καλωσορίζω φυσικά την επέκταση ε, του κανονισμού και στον τομέα αυτό, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ ε, προσεκτικά τι θα ενταχθεί εκεί και τι δεν θα ενταχθεί. Για να το πω, μα ε, κανείς δεν θα προσπαθήσει να ξεπλύνει χρήματα ε, στη ε, κρατική λαχιοφόρο αγορά γιατί οι πιθανότητες είναι 1 προς 1,3 εκατομμύρια ε, ε, ότι θα είναι ξέπλυμα. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ποια είναι εκείνα τα τυχερά παιχνίδια και ποιο λόγο προσφέρεται για νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων και όχι ε, τα επίσημα κρατικά λαχεία. Ε, και επίσης ε, και κατά την καταπολέμηση φορολογικού εγκλήματος είναι κάτι που μα ενδιαφέρει πολύ. Ευχαριστώ. On behalf of the EPP, I give the word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 να αντιληφθούμε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για την νομιμοποίηση. Μπαίνει χρήμα στην αγορά και νομιμοποιείται. Αυτό το φαινόμενο ε, έχει αυξανόμενη σημασία τα τελευταία χρόνια και ε, συνιστά μεγάλο κίνδυνο για την πραγματική οικονομία. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο το ζήτημα της νομιμοποίησης εσόδων. Ορισμένες φορές αναλαμβάνεται δράση σε πολλά μέρη ταυτόχρονα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διευρύνει το πεδίο των υφιστάμενων διατάξεων από όλους τους εμπλεκόμενους, τουλάχιστον ένας βρίσκεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν κάνει κάποιος μια χρηματική συναλλαγή πρέπει να δίνει και κάποιες πληροφορίες. Προβλέπει ο κανονισμός ότι θα πρέπει να δοθεί ο αριθμός ε, ταυτότητας ε, του δικαιούχου καθώς και του ε, ατόμου που κάνει το έμβασμα. Στη συνέχεια αποθηκεύονται τα στοιχεία για ελάχιστο διάστημα 5 ετών. Σε περίπτωση παραβίασης κανόνων προβλέπονται κυρώσεις που ανέρχονται ως και σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Ή στο 10% του κύκλου εργασιών. Η αξιόπινη πράξη του, της νομιμοποίησης ε, παρανόμων εσόδων υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ε, φυσιολογική συμπεριφορά των νομοταγών πολιτών. Ε, είναι σίγουρο ότι αν συλλέξουμε χρήματα από ανάκτηση τέτοιων εσόδων θα χρηματοδοτήσουμε την δράση καταπολέμησης αυτού του φαινομένου. Όμως πρέπει να είμαστε λογικοί για να είναι αναλογική η δράση μας ως προς ε, τους στόχους που έχουμε θέσει. Πιστεύω ότι οι δράσεις που αναλαμβάνουμε δεν πρέπει να συνιστούν ε, ε κόλλημα για όλους όσους ε, εργάζονται σε αυτόν τον τομέα ή επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ε, το σύστημα μεταφοράς κονδύλιων. Δεν πρέπει να διώξουμε με αυτές τις νέες διατάξεις από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους ε, νόμιμους ε, πληρωτές και δικαιούχους. Ε, εξάλλου η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου συνεπάγεται ένα κόστος το οποίο μετακυλίεται στους πελάτες. Τα δεδομένα δε που αποδικεύονται έχουν ευαίσθητο χαρακτήρα και άρα θα πρέπει κάποια δημόσια αρχή να ελέγχει τον οργανισμό που αποθηκεύει αυτά τα στοιχεία. Δεν προβλέπεται όμως αυτό στην πρόταση κανονισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και να οριοθετήσουμε τη δράση μας. Δηλαδή, για ποιους σκοπούς είναι δυνατή η χρήση αυτών των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων και ε, να χρησιμοποιηθεί για έκνομους σκοπούς ε, αυτή η βάση δεδομένων. Εξάλλου στο άρθρο 114 συνθήκες Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, που είναι κοινομική βάση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας διαβλέπω κάποια προβλήματα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ε, βασιστούμε μάλλον στο άρθρο 352 και στη ρήτρα ευελιξία ε, που υπάρχει εκεί. Για το πεδίο εφαρμογή. μιλάμε για συλλογή προσωπικών δομένων από τους διαμεσολαβητέ, εκ των οποίων ο ένα τουλάχιστον πρέπει οπωσδήποτε να είναι στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογή τη πρόταση. Θυμάμαι και τι συζητήσει μα ε, για το φόρο επιχρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Λοιπόν, η ηθαγένεια θα πρέπει να είναι το κριτήριο, ώστε να καταστεί κάποιο επιλέξιμος για τη συλλογή ε, προσωπικών δεδομένων για μια χρηματοπιστωτική συναλλαγή μεταξύ δύο πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει η χώρα εκτός αυτής. Είναι ίσως λίγο ε, υπερβολικά αυτά τα σενάρια που σας εκθέτω, αλλά έχω σοβαρούς ενδιασμούς και περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω την υπόλοιπη συζήτηση. Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Νίτρας. Από πλευρά των πρασίνων δεν θέλετε το λόγο. Ω, συγγνώμη, φιλελεύθερος. Ξέχασα τους φιλελεύθερους, έγινε και η Σοφή εδώ. Mm. Ζητώ συγγνώμη, τα έχω χαμένα. Ναι. Ο κύριος Τόρβαλ θα πάρει πρώτος το λόγο, γιατί αφήστε που έχει δικαίωμα, έχει ζητήσει κιόλας το, το λόγο. Θα μιλήσει εξ ονόματος των φιλελευθένων. Ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε μια έρευνα που έγινε από τα Ηνωμένα Έθνη για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ περνάνε μέσω από την νομοποίηση εισόδων παράνομες δραστηριότητες. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 2,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Λιγότερο από 0,2% των πόρων αυτών επαναπατρίζονται Καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αυτά είναι απλές εκτιμήσεις. Τα οριστικά στατιστικά δεδομένα ενδεχομένω είναι αδύνατο ποτέ να διατεθούν. Αυτό το οποίο μας λένε όμως τα στοιχεία αυτά είναι ότι η νομοποίηση εσόρων παράνομων δραστηριοτήτων είναι ένα διεθνές διασυνοριακό πρόβλημα. Ξέρετε ότι η νέα τεχνολογία με τις συνθήκες εσωτερικής αγοράς δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες ε, για νομοποίηση εισόδων παράνομες δραστηριότητες και επομένως περισσότερες προκλήσεις για την καταπολέμησή της. Απαιτείται λοιπόν να υφίστανται διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα αυτό είναι διασυνοριακό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα και συνέπεια ανάμεσα στους εθνικούς κανόνες και θα πρέπει το νέο αυτό νομοθέτημα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Χαιρετίζω λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας, ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να θίξουμε. Πρώτον, η επέκταξη του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία σημαίνει ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία και αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη, ιδίω στα κράτη-μέλη εκείνα όπου δημόσιοι φορεί εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και με τη σειρά του κατά αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούν στα εξωτικά ταμεία. Είναι πολύ σημαντικό η νέα αυτή διάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην δημιουργήσει επιπλέον γραφειοκρατικό άκθος για αυτές τις χώρες. Όσον αφορά τώρα την ταυτοποίηση των ε, πελατών για τα τυχερά αυτά παιχνίδια, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, ο κύριος Τόλβατς, ευχαριστούμε μάλλον. Η κυρία Ντιβέλτορ θα έχει το λόγο. Και συνέχεια ο κύριος Γίγκελ. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε και εμεί υπέρ τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν από του προλαλήσαντε. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να προσθέσουμε κάποια επιπλέον σημεία. Πρώτον, πιστεύω στεναρά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εντοπίσουμε ποιο είναι ο πραγματικό οικονομικό δικαιούχο. Με ποιον συναλλάσσεται δηλαδή μια επιχείρηση και νομίζω ότι στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου θα μπορούσαμε να προβλέψουμε πάρα πολλά πράγματα. Η ουσία όμως είναι να εφαρμόζεται στη συνέχεια το κοινοτικό δίκαιο. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι να επιμείνουμε στο ζήτημα της εφαρμογής, της επιτόπιλοποίησης και όχι απλώ το τι λέμε εμεί θεωρητικά εδώ στι Βρυξέλλε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμείνουμε στο ζήτημα τη εφαρμογή. Και δεν αρκεί να καταστήσουμε την οδηγία πιο αυστηρή, ή να καταλήξουμε σε έναν κανονισμό. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μηχανισμούς βάσει των οποίων θα μπορούμε να βλέπουμε αν οι υφιστάμενοι κανόνες όντως ισχύουν. Πρόσφατα στην Κύπρο είδαμε πως ε, εκδηλώθηκε το πρόβλημα αυτό. Επίσης, η δημιουργία ενός μητρώου που θα περιλαμβάνει όλες τις υπόχρεες οντότητες, δηλαδή ακόμα και τα διαπιστεύματα, καταπιστεύματα, με συγχωρείτε, είναι κάτι πολύ σημαντικό και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε περισσότερη διαφάνεια στο ζήτημα του οικονομικού δικαιούχου. Επίσης, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην εσωτερική αγορά να γνωρίζει ακριβώς με ποιον συναλλάσσεται και να μην έχει απλώς τον αριθμό ενός ε, γραμματοκιβωτίου κάπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το όνομα της επιχείρησης, την ταυτότητα της επιχείρησης. Σαφώς αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε κάποιους ε, κινδύνους, σε κάποια προβλήματα. Ο κύριος Κάριν αναφέρθηκε και σε αυτή τη διάσταση, αλλά θεωρώ ότι ε, στα πλαίσια μιας οικονομίας αγοράς είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς με ποιον συνεργάζεται. Και δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δημιουργούνται όλο και περισσότερες δυνατότητες για κάποιες επιχειρήσεις να μην αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα των τυχερών παιχνιδιών τα όσα προβλέπονται εδώ πέρα δεν είναι απόλυτα συνεπή με τα όσα ισχύουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τις νέες αυτές προτάσεις. Ουσιαστικά το πρόβλημα να έγκυται περισσότερο στα τυχερά παιχνίδια online, στα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια. Ίσως εκεί πέρα να πρέπει να αστιαστούμε περισσότερο. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι στη Γερμανία υπάρχουν κάποια προβλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην πραγματική οικονομία, όχι μόνο ε, στην επιγραμμική οικονομία ή στις πραγματικές υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και όχι μόνο σε αυτές οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να κάνουμε μία διάκριση και να δούμε ακριβώς που έγκυται ο κίνδυνος και να μην επιβαρύνουμε τελικά τους τομείς εκείνους στους οποίους δεν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε πού έχουμε παράνομες δραστηριότητες, πού έχουμε εγκληματικότητα και πού όχι. Αυτό το οποίο βλέπω όμως στη Γερμανία είναι ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εγκληματικής δραστηριότητας και εκτός εικονικού ηλεκτρονικού κόσμου. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, το γεγον... για τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών νομισμάτων. Νομίζω ότι δημιουργείται πρόβλημα πολλές φορές από το γεγονός ότι ορισμένες χώρες επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση τόσο του πραγματικού νομίσματος όσο και ενός εικονικού νομίσματος για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. και σε ορισμένε περιπτώσεις έχουμε δει ότι σε κάποιες περιφέρειες χρησιμοποιούνται ακόμα και κάποιες ε, περιφερειακές οικονομικές μονάδες, κάποια περιφερειακά οικονομικά νομίσματα. Και σε ορισμένε περιπτώσεις ανακαλύπτουμε ότι πίσω από τη χρησιμοποίηση αυτών των ε, μονάδων μέτρησης κρύβονται ολόκληρα σχέδια παράνομων οικονομικών δραστηριότητων. δραστηριοτήτων. Με συγχωρείτε. Και ποιο λόγο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ασχοληθεί και με το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ενδεχομένως ως προς αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί και η πρόταση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον όντως έχουμε δει κάποια τεράστια σκάνδαλα να διεξάγονται σε κάποιες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι θα μπορούσε επίσης να ενδυναμωθεί και ο ρόλος του ευρωπαϊκού επόπτη και τέλος θα ήθελα σας πω ότι το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε μια πραγματική εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντεξάγουμε συζητήσεις με τα κράτη-μέλη για πίνακες συγκρίσεων που θεωρούν ότι πάρα πολλές φορές ε, είναι κάτι το οποίο βαρύνει ιδιαίτερα την ε, γραφειοκρατία στα κράτη αυτά, αν δεν εφαρμόζεται στη συνέχεια στην πράξη η οδηγία και ο κανονισμός. Στην ε, χώρα που γνωρίζω καλύτερα, την Γερμανία, ξέρω ότι έχουμε αρκετές περιπτώσεις νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το επίπεδο συμμόρφωσης με τους κανονισμούς είναι χαμηλό και θεωρώ ότι με τις νέες αυτές προτάσεις θα καταφέρουμε να έχουμε τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια καλύτερη συμμόρφωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το φαινόμενο της μη εφαρμογής των ε, κοινοτικών διατάξεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα είναι συντηρητική ο Ντέρκ, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Θα διαβάσω τη δήλωση κυρίας Κράτσα που δεν μπορούσε να έρθει καλωσορίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, χρήματος. Ε, αυτή η δραστηριότητα και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ενέχει αξιόπινες πράξεις που πρέπει να κατασταλούν με αυστηρό τρόπο σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με όλα τα κατάλληλα μέσα. Τονίζει την ανάγκη επίση για τις ανεπτυγμένες χώρες να συνασπιστούν και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία ειδικότερα ε, στις εισαγωγικές του παρατηρήσεις ε, τονίζει ότι αναμένει από το σχέδιο της ΕΚΟΝ να τονίσει την ανάγκη για τα κράτη-μέλη ε, να μεταφέρουν γέρος και δεόντος στην εθνική νομοθεσία τους όλα τα διεθνή πρότυπα για τη χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για το ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότης τρομοκρατίας. αν δεν είναι βέλτιστη η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία αυτού του νομοθετήματος, αυτό θα αποτελέσει κόλλημα στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κίνδυνο για την συνοχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θεωρεί ότι είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε τα περί, τις απαιτήσεις περί δέουσας επιμέλειας για τους, κατα, για τους πελάτες και τους πραγματικούς δικαιώχους σε σχέση με τη συμπερίληψη των ε, παρόχων ε, για τα τυχερά παιχνίδια θεωρεί ότι πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά αυτή την ιδέα διότι ε, έχει τόσες πολλές ε, αρνητικές ε, ιονίες επιπτώσεις αυτό το φαινόμενο που χρειάζεται στενή παρακολούθηση για τους εθνικούς λαχνούς, δε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ε, θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πεδίο της νέας πρότασης για τη μείωση από τους 15.000 σε 7.000 για τις εμπορικές συναλλαγές. Ε, πιστεύει ότι χρειάζονται προληπτικά μέτρα και αν εγκριθεί τελικά αυτό το κατόφλι θα πρέπει να ισχύσει μόνο για οικονομικές συναλλαγές. Ο κύριος Στρέτσεκ ε, τονίζει επίσης ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης θα ενθαρρυνθούν για να συμμορφωθούν με τις νέες διατάξεις. Αυτά τα πάω όλα. Ευχαριστώ. Mm. θα ήθελε κάποιος άλλος ε, να πάρει το λόγο που δεν τον προσέξαμε από την ΚΟΕ. Έχω και εγώ διάφορα να πω και ζητώ συγγνώμη που έχασα ένα τμήμα της συζήτησης γιατί επίκειται δύσκολη ψηφοφορία, είχαμε θέματα με τον κατάλογο. Νομίζω ότι είναι επίκαιρη η αναθεώρηση της οδηγίας ε, για το ξέπλυμα χρήματος. Έχουμε τις συστάσεις ε, τις περσινές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην εξετάσουμε μόνο αυτή, αυτό το νομοθέτημα, διότι η επιθετική φοροδιαφυγή, πολλαπλασιασμό των φορολογικών παραδείσων, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και παρανόμηση εσόδων είναι τμήματα του ίδιου παζλ. Ε, όπως είπαν και άλλοι, ε, πρέπει να ξέρουμε βασικά ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι. Beneficial beneficial owners. Ε, αυτό συζητείται τώρα από την ομάδα G8 και νομίζω ότι σε λίγες ημέρες θα ξέρουμε περισσότερα για αυτό το ζήτημα. Θα ενισχυθούν ε, τα εθνικά συστήματα, νομίζω ούτως ή άλλως. Κάτι άλλο που σχολίασαν οι συναδέλφοι είναι για τα τυχερά παιχνίδια. Αν πρέπει ε, να ε, τεντώσουμε κι άλλο την οδηγία για να καλύψουμε κι άλλους τομείς. Ας μην φοβούμαστε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής στο μέτρο του δυνατού, ενδεχομένως να ανακύψει ένα θέμα αναλογικότητας βεβαίως. Γιατί όπως φαντάζεστε διάφοροι κανονισμοί ε, καλύπτουν έναν εθνικό λαχνό, παραδείγματος χάρη ένα εθνικό σύστημα στοιχημάτων και αυτό ίσως ε, επειδή αυτό σχετίζεται περισσότερο με μικρές τοπικές οργανώσεις. Άρα πρέπει να εξετάσουμε αν είναι αρκούντως αναλογικές οι προτάσεις ε, προτού σπεύσουμε να αποφασίσουμε αν κάτι θα συμπεριληφθεί ή όχι. Αυτά είχα να πω. Απ και κάποιος άλλος θέλει το λόγο, ο Ρουί Ταβάρης. Κανένα πρόβλημα δεν είναι το ταμπελάκι μου εδώ, δεν λέγομαι Λάμπερ, βάρες λέγομαι. Ε, να σας πω ότι παρακολουθώ τις εξελίξεις αυτού του φακέλου ε, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ε, είμαι νέος αναπληρωτής ε, εδώ στην ΕΚΟΝ ε, για την Ειδική Επιτροπή ΚΡΙΜ, ξέρετε, προετοιμάσαμε μια θεματική μελέτη για την φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα και το οργανωμένο έγκλημα. Και εκεί υπάρχουν κάποιες ε, ενδιαφέρουσες ιδέες για τον εντοπισμό των δικαιούχων και για τη δέουσα επιμέλεια των τραπεζών για να ε, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου όταν κάποιος από τον κατάλογο των πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων ε, εμπλέκεται στην ε, συναλλαγή. Έχουμε και την ε, ΦΑΤΦΕ, την ειδική δράση χρηματοοικονομικής δράσης, αλλά αυτά τα είπαν οι συνάδελφοι. Λοιπόν, σε συνδυασμό με αυτή τη μελέτη της ειδική υποεπιτροπής ΚΡΙΜ, ε, μπορούμε να υποφεληθούμε από τα θεματικά έγγραφα. Θα τα στείλω και στους ε, εισηγητές και στους κοιόδης και στη γραμματεία αν το επιθυμείτε γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ιδέες. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ο Κρισιανής Κάρενς. Ευχαριστώ πολύ. Από όλα τα σχόλια φαίνεται ότι βρισκόμαστε όλοι περίπου στο ίδιο πνεύμα. Οι περισσότεροι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ανάγκη να εξακριβώνεται ο τελικός δικαιούχος και πολύ επίσης, όπως και η πρόεδρος, αναρωτήθηκαν τι γίνεται με τα τυχερά παιχνίδια και αναλογικά πώς και συμμετέχει και τι σχέση υπάρχει με τα κρατικά λαχεία, ε, αν είναι κάποιος ιδιωτική επιχείρηση στοιχημάτων ή τυχερών παιχνίων. Προφανώς ο κίνδυνος δεν είναι να ξεπλένει κάποιος χρήματα στα κρατικά λαχεία, αλλά αλλού. Αν σκεφτώ, ας πούμε, τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου δεν είναι τα κρατικά λαχεία. Οι εθνικοί φορείς... Ε, θα συνεργαστώ με τους υπολείπους και οδησηγητές ε, και την άλλη έκθεση για τον κανονισμό και ελπίζω και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε κάπως να ε, βελτιώσουμε και να ε, διευκρινίσουμε λίγο, να αφενήσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Πρόεδρος, η Κομισιόν παρίσταται, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Και καλό θα ήταν να τις ακούσουμε, ε, να δούμε αν σημειώνουν τα όσα τους προτείνουμε. Γιατί ακούσαμε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια αιτήματα να απευθύνονται. Έχουμε και άλλο συγκητή. Ναι, να δώσω το χρόνο μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει η κυρία Κλέβα. Α, εσείς θέλετε να την ακούσετε οπωσδήποτε την Επιτροπή. Καλά. Η συγκήτρια της Επιτροπής Λίμπε προτιμά να δώσει το χρόνο της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Thank you very much, Mrs. Uh, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη δυνατότητα που μας δίνετε. Θα απαντήσω λοιπόν καταρχάς στα ερωτήματά σας. Δεν θα ξεκινήσω με τα πιο πολύπλοκα ζητήματα. Πρέπει απλώς να σας πω ότι αναφερθήκατε αρκετά στο εξή ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν αναφερόμαστε περισσότερο στις πληροφορίες όσον αφορά σε ποιον πηγαίνουν τα χρήματα, όσον αφορά τον δικαιούχο. Μα έχουμε ήδη το σύστημα ΣΥΠΕ, το οποίο μας επιτρέπει πραγματικά να έχουμε την απαραίτητη χνηλασιμότητα τόσο για τον πληρωτή όσο και για τον δικαιούχο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να συμπεριλάβουμε συγκεκριμένε πληροφορίε όσον αφορά τον δικαιούχο για ένα έμβασμα. Υποτίθεται ότι η πληροφορία αυτή υπάρχει και την πληροφορία αυτή την έχει η τράπεζα. Το άλλο ερώτημα το οποίο θέσατε έχει να κάνει με τις δυσκολίες τις οποίες έγκυται για κάποιες μικρές οντότητες και αναφέρεστε εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, σε δικηγόρους. Πρέπει να σας πω ότι εδώ πέρα αναφερόμαστε όμως μόνο σε τράπεζες και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία κάνουν εμβάσματα. Επομένω, τα νομοθετήματα εδώ πέρα δεν αναφέρονται σε μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και οντότητες. Επίσης είπατε τι διαφορές μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στην ΣΕΠΑ, την οδηγία για τις χρηματοπιστωτικές πληρωμές ε, με τους συναδέλφους μου που εργάζονται για τα ζητήματα αυτά έχω συζητήσει και πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαφορές και αποκλήσεις. Αν εσείς ε, έχετε εντοπίσει κάποιες αντιθέσεις, κάποιες διαφορές, τότε ας μας το πείτε για να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τα σημεία αυτά. Να αναφερθώ και σε κάποια άλλα ζητήματα με την άδειά σα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε ένα ζήτημα το οποίο ακούστηκε πάρα πολλές φορές, τυχερά παιχνίδια το γεγονός ότι δεν μπορούν να καλυφθούν κάποιες κρατικές λαχιοφόρες ε, αγορές. Πολλά κράτη-μέλη πιστεύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια για να νομοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες δεν διεξάγεται με τον τρόπο τον οποίο αναφέρατε εσείς εδώ πέρα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι ευφυείς τρόποι προκειμένου να νομοποιήσει κανείς ε, έσοδα από παράνομες δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από την οδηγία. Έχουμε επίσης και το κατόφλι των 2.000 ευρώ. Ξέρετε ότι ήδη υπάρχει λοιπόν το ζήτημα αυτό της αναλογικότητας. Θέτουμε ένα κατόφλι 2.000 ευρώ. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Γκίγκελς ε, για το Liberty Reserve, δεν προβλέπεται εδώ πέρα μία ρύθμιση για, τις, για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εξετάσαμε πάντως το ζήτημα αυτό πάρα πολύ προσεκτικά και μέχρι στιγμής δεν καλύπτονται από, το από το καονιστικό αυτό πλαίσιο. Το έχει εξετάσει πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχει να κάνει μόνο με την νομοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θέλουμε να δούμε αν δικαιολογείται από αναλογικής πλευράς να εντάξουμε στον κανονισμό αυτό και την περίπτωση στην οποία αναφερθήκατε. Αυτά μπορώ να σας πω μέχρι στιγμής. Δεν είχαμε και πάρα πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και επίσης σας ευχαριστώ, ε, κυρία Κλέβα, που δώσατε το χρόνο σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας παρακαλώ. Ξέρω ότι έχουμε ψηφοφορίες, αλλά δεν ακούω ότι τον ίδιο μου τον εαυτό θα μιλάω. Λοιπόν, μέχρι να ησυχάσετε δεν θα γίνει τίποτα. Okay, I think um, everybody should... Λοιπόν, έχετε όλοι το κατάλογο ψηφοφορία σας. Γιατί μπορεί να είναι λίγο σφιχτές οι ψηφοφορίες. Ας κάνουμε λοιπόν μια δοκιμαστική τώρα παρακαλώ, ηλεκτρονική δοκιμαστική ψηφοφορία. You have your group voting list? No. You want to vote? I'll have to try and follow them. At the moment we've only got 39 members here. Λοιπόν, έχουμε 39 μέλη και μόνο 33 ψήφισαν για τη δοκιμαστική. 35 have pressed button. 35 40 είναι συνδεδεμένοι, 38 ψηφίζουν Πλάκα έχει να τα παρακολουθείς αυτά. 41 συνδεδεμένοι, 40 ψήφισαν. Πάντα ένας έχει βάλει κάρτα αλλά δεν ψηφίζει. Γιατί μήπως δεν δουλεύει το μηχάνημα ή κάποιος έτσι αντιδραστικά επίτηδες το κάνει. Okay, there's a card plugged in that hasn't voted. There are now two cards. Λοιπόν, ψήφισαν 40, 42 κάρτες. 41 έχει έχουν ψηφίσει. Παραμένει μία κάρτα στο μηχάνημα που δεν ψηφίζει. Εντάξει, λοιπόν, αρχίζουμε. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Άννης Ποδηματά, θέσπιση ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Παρακαλώ να σταματήσουν οι ιδιωτικέ συνομιλίες, γιατί η αίθουσα είναι τέτοια που όταν μιλάτε εγώ δεν ακούω τίποτα. And if you're talking, I'm going to stop. Και όποτε μιλάτε θα σταματάω, οπότε θα ψηφίζουμε για ώρες. Αυτό ισχύει και για το προσωπικό και όλους τους υπολείπους επισκέπτες και παρατηρητές. Δεν ακούω ούτε τον εαυτό μου. Σας παρακαλώ μην μιλάτε, είναι η αίθουσα τέτοια. Λοιπόν, ωραία. Η τροπολογία υπάρχει 21 και 22 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 23 Επέ. κατά αποχές απορρίπτεται. 24 Επέ. κατά αποχές. Καλύτερα να την ελέγξουμε παρακαλώ. Εγκρίνεται 25 υπέρ, 17 κατά. Η τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 70 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 τι θα ψηφίσεις και άλλαξε θέση. Λοιπόν, 18 υπέρ, 24 κατά απορρίπτεται η τροπολογία. Η τροπολογία 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G προφορική τροπολογία λέει εδώ η πράσινη. Οι πράσινοι έχουν μια προφορική τροπολογία. Θα ψηφίσουμε πρώτα την προφορική και μετά τον συμβιβασμό όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ λοιπόν της προφορικής τροπολογίας. Κατά αποχές έλεγχο χρειάζεται αυτό. Είναι μόνο η προφορική τροπολογία αυτό που ψηφίζουμε. Okay. Rachel. Okay. Votes. Right, we're closing the vote. Τι ψηφίζεις υπέρ κατά 21 υπέρ 20 κατά εγκρίνεται. in Ναι, έχουμε μία ψήφο κατά, λέει η κυρία ε, Ματίας είναι υπέρ. Δεν θέλω να ακούω τι ώρα κοιμηθήκατε. Τι ήταν αυτά, τρεις η ώρα κοιμήθηκα. Λοιπόν, ε, ήρθαν δύο, μία υπέρ, μία κατά. Άρα κερδίζει με μία ψήφο διαφορά. Και ψηφίζουμε το συμβιβασμό όπως τροποποιήθηκε με την προφορική. Ε, λοιπόν, συμβιβασμός όπως τροποποιήθηκε ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτός αν θέλει κανείς να το ελέγξουμε. Όχι. Η τροπολογία 100 είπε. Κατά. Άποχες. Αυτό θέλει έλεγχο όμως. Right, 100. Η τροπολογία παριθμών 100. Η Αρλίν έχει ένα πρόβλημα με την κάρτα της. Ψηφίστε τώρα, δύο δεν έχετε ψηφίσει ακόμα βλέπει τα φώτα να ανάβουνε. Δουλεύουν όλες οι κάρτες. Okay, right, votes closed. περας ψηφοφορίας εγκρίνεται 24-18. Συμβαστική H. Έχουμε μια καθυστερημένη προφορική τροπολογία των φιλελευθέρων για την εξαίρεση για τα συνταξιοδοτικά ταμεία pension funds. Το ίδιο ισχύει και για κάποια άλλα τμήματα. Η Ποδηματά, παρακαλώ. Yes, Sharon, thank you. I... Ευχαριστώ, Σάρον. Θέλω να τονίσω ότι δεν καταλαβαίνω αυτήν την προφορική τροπολογία. Κάναμε πάρα πολύ μακρές συζητήσεις μέχρι αργά χτες το βράδυ, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και ε, καλύψαμε και το ζήτημα των συνταξιοδοτικών. Οπότε δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτή την, ε, το αίτημα τελευταία στιγμής για την εξαίρεσή τους. Does anybody from, from... Θέλει κάποιος από τους φιλελεύθερους ή να ψηφίσουμε απλώς. Λοιπόν, ξέρω ότι τρεις μπορούν να προβάλλουν ενστάση, αλλά τείνουμε να μην το κάνουμε ένα στον άλλον αυτό για προφορικές τροπολογίες. Ε, η γενική τάση είναι να λέμε άντα, ψηφίσουμε τότε. Ε, είναι λιγότερο επιθετικό, καταλαβαίνετε, το να ψηφίσουμε. λεπτάκι. Ναι, Ραμόν. Θέλω να εξηγήσω, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, διαπραγματευόμασταν μέχρι τελευταία στιγμή. Εγώ ήμουν ε, τα τελευταία χρόνια επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για την ομάδα μου και μου ζητούσαν να χαρακτηρίζουμε από συνέπεια στη δράση μου, αλλά θέλανε ταυτόχρονα να περάσουν και ένα πολιτικό μήνυμα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν ενστάσεις για αυτή την προφορική τροπολογία ή όχι. Πρόεδρος, εγώ νομίζω ότι θα ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία και μετά ε, θα ψηφίσουμε για τη συμβαστική. Με ή χωρίς. Λοιπόν, ας αρχίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η προφορική τροπολογία. Τώρα συμβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συγγνώμη, να το ελέγξω. Συμβαστική H. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 33 ψήφοι υπέρ 10 κατά. Εγκρίνεται. On page It's on page I Στη σελίδα 7. Τη δικιά μου 7. Η 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί με δυσκολεύει αυτή η αίθουσα δεν βλέπω καλά. Ψήφισαν όλοι. Votes closed. Πέρας. Εγκρίνεται 24 προς 19. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με τον ίδιο αριθμό ψήφων. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 134 ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ ένα λεπτάκι και έκανα λάθος καταπίπτει οι 147 και 149 και 17 καταπίπτουν και φτάνουμε στην 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 budget υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 155 υπέρ κατά έλεγχος, έλεγχος 155 παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας, εγκρίνεται 23 ψήφοι προς 21. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 Ψήφισαν όλοι. Άλλη μία ψήφο θέλω. Πέρας. Εγκρίθηκε 27 προς 17. 170 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική α σε διάφορα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα συμβαστική βήτα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. 30. Έλεγχος για 30. Πέρας. 27 ψήφι προς 18 εγκρίθηκε όντως. 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Α, ναι, η συμβαστική C. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι αυτή συγκαλύπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 53 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 54 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 55 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλά, ένα λεπτάκι. Είναι ταυτόσιμη. Την καλύψαμε με τη συμβαστική δέλτα. H, συγγνώμη. Την 57 ξανά, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά. Κατέπεσε 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του τροποποιηθέντος κειμένου ηλεκτρονική ψηφοφορία. 30 ψήφοι υπέρ, 12 κατά και 3 αποχές. Και τώρα ψηφίζουμε για το νομοθετικό ψήφισμα. Λείπουν δύο. Πέρας. 30 προς 10 και 4 εποχές. Άννη θέλεις τον λόγο. Ευχαριστώ Σάρον. Θέλω να ευχαριστήσω τους Κιώδης, κυρίως τον Όντμαρ Καρές Δραμοραμόζα, Φίλιπ Ραμπέτς και Μαρίζα Ματίας για την ε, ε, αξιόλογη συμβολή τους. Τονίζω ότι με δεδομένη τωρινή κατάσταση και το έντονο λόμπινγκ από τη βιομηχανία για να δολοφονήσουν τον νεοφόρο, ε, ήταν απαραίτητη η δέσμευση και η προσήλωση των συναδέλφων για να καταλήξουμε σε αυτό το συμβιβασμό. Χάρη στη δέσμευση και αφοσίωσή τους εγκρίνουμε σήμερα στην ΕΚΟΝ μια θέση που ε, στοιχειοθετεί και αποδεικνύει την συνέπεια και την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σάρον Μπόλς ήθιστε να δίνουμε στον εισηγητή το λόγο, ε, στους κοιόδης πάλι όχι. Όλοι θέλουν τα 15 λεπτά δημοσιότητας, αλλά εμείς δεν προλαβαίνουμε. Περνάμε στο σημείο 8 για την ε, ψηφοφορία για τον τραπεζικό τομέα και τη μεταρρύθμιση του. Okay, Ας περάσουμε τώρα στην έκθεση της Αρλίν για τη διάρθρωση του τραπεζικού τομέα και η Αρλίν Μακάρθη μου ζήτησε το λόγο τώρα στην αρχή πριν την ψηφοφορία και όχι στο τέλος γιατί θέλει να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Επομένως έχει το λόγο. Δεν έχω να πω σπουδαία πράγματα. Ήθελα απλώ να μιλήσω εκ των προτέρων γιατί νομίζω ότι θα έχετε δει ότι υπάρχουν περίπου 400 τροπολογίες και με τους κοιόδης ηγητές καταφέραμε να συνεργαστούμε ιδιαίτερα επικοδομητικά και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης ε, εισηγητές για την επικοδομητική, αποτελεσματική και γρήγορη αυτή συνεργασία. Επιφέραμε πολύ σημαντικές αλλαγές γιατί εν τέλει υπήρχαν πολλοί που δεν θέλαν να ασχοληθούν με τις διάφορες λεπτομέρειες αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας, θέλαν να βασιστούν κάπως σε κάποιες βασικές αρχές και δεν θέλανε να επισέλθουν σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και είπαν ότι αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει στα πλαίσια μιας ευρύτερης συζήτησης που θα πρέπει να γίνει για μια πραγματική νομοθετική πρόταση. Ελπίζω λοιπόν να δεχτείτε την προσέγγιση αυτή. Σα άκουσα ω ηγητέ, έκανα και ίδια κάποιε αλλαγέ, τι οποίε δεν επιθυμούσα αρχικά να κάνω, αλλά για λόγου συμβιβασμού και συνένεση το έκανα αυτό και ελπίζω εν γέννη ότι είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Και κατά αυτόν τον τρόπο καταφέραμε τελικά να καταλήξουμε σε κάποιε συμβαστικέ λύσει και να μειώσουμε τον αριθμό των αρχικών τροπολογιών. Σάρων, στα επιμέρου σημεία θα ζητήσω το λόγο εφόσον χρειάζεται για να δώσω περαιτέρω εξηγήσει κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία δηλαδή, πρόεδρο. Όντω υπάρχει ένα τομέα όπου υπάρχει μια κάποια σύγχυση για το τι είναι συμβατό και τι όχι στι προτινόμενε τροπολογίε. Θα καταφέ... Πιστεύω θα καταφέρουμε όμω να βρούμε μια λύση. Ε, εντοπίζεται αυτό στην αιτιολογική σκέψη, θα ψηφίσουμε για τι αιτιολογικέ σκέψει. Α ξεκινήσουμε πάντω με τη συμβαστική α υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Γ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική D, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική η, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H. Έχουμε δύο προφορικές τροπολογίες και μία χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Θα γίνει ψηφοφορία με την σειρά που τη βλέπετε εδώ πέρα στον κατάλογο ψηφοφορίας, καταρχάς οι προφορικές τροπολογίες από το ΕΛΚ, προφορική τροπολογία του ΕΛΚ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία των φιλελευθέρων, συγγνώμη, με συγχωρείτε παρακαλώ. Με κατά της προφορικής τροπολογίας των φιλελευθέρων, υπάρχει κάποιος άλλος που είναι κατά. Μάλιστα, λοιπόν, δεν θα ψηφίσουμε τότε αυτή τη φορά όπως κάνουμε συνήθως. Λυπάμαι βέβαια για κάτι τέτοιο, για αυτό το οποίο συνέβη. Επομένως, στο πρώτο τμήμα ήταν οι προφορικές τροπολογίες, μάλιστα. Θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα που περιλαμβάνει την προφορική τροπολογία του ΕΛΚ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία I υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική L σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 396 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 394 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος για την 394. Υπάρχει ένα, μία επιπλέον ψήφος από τους σοσιαλιστές. Όλα εντάξει τώρα. 26 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στο αρχικό κείμενο. Μάλλον δεν ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Πάμε στην παράγραφο 18, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 398 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 398. Πέρας. Απορρίπτεται 21 ψήφος, ψήφι 24 κατά. Τροπολογία 401 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 401. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 401. Ψηφίσατε όλοι, εγκρίνεται, 27 υπέρ 18 κατά. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 405 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση και την 405 σας παρακαλώ. Ταυτόσημη με την 406 υπέρ, ε, μάλλον συγγνώμη, πέρας Απορρίπτεται. 22 υπέρ, 23 κατά. Περνάμε στη 410 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική M σε τέσσερα τμήματα. Εγώ τουλάχιστον βλέπω τέσσερα τμήματα. Σε τέσσερα τμήματα λοιπόν συμβαστική αίμα απόλυτα ξεκάθαρα τα πράγματα όσον αφορά αυτή τη συμβαστική τροπολογία. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τα πράγματα με κάποιο ξεκάθαρο τμήμα. Στο πρώτο τμήμα λέμε ότι ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιλάβει διατάξεις προκειμένου να ενισχυθεί η ε, προσωπική λογοδοσία και ευθύνη όσον αφορά τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και των ε, ξεχωριστών οντοτήτων σε επίπεδο μήλου. Στο τμήμα 2 αναφερόμαστε στο ίδιο κείμενο, χωρίς όμως τη φράση «in the separated entities and at group level». Συγγνώμη, δεν παρουσιάζεται πολύ καλά αυτή η συμβαστική τροπολογία στο έγγραφο και στο τρίτο τμήμα τι γίνεται. Έχουμε τρία τμήματα λοιπόν, τρία τμήματα, κατάλαβα μάλιστα. Στο πρώτο τμήμα καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει διατάξεις προκειμένου να αυξηθεί η προσωπική ευθύνη και λογοδοσία των μελών Διοικητικών Συμβουλίων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έπειτα στο δεύτερο τμήμα έχουμε το in the separate entities and at group level υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στο τρίτο τμήμα, πρώην τέταρτο, προτείνεται στο περιβάλλον αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει και το καθεξής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Α, το ΕΛΚ άλλαξε άποψη. Συγγνώμη. Ένα λεπτό, ησυχία παρακαλώ. Εκτός μικροφώνη παρέμβαση. Ε, θα κάνουμε πρώτα μια ηλεκτρονική επαλήθευση των όσων προτείνονται εδώ στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ο κύριος Γκοζές, πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα αν δεν ησυχάσετε και πρέπει να καταφέρουμε να ακούμε και τους συναδέλφους και να μπορώ και ίδια να μιλήσω προτείνεται ότι στο περιβάλλον αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει πώς μπορεί να ενθαρρύνει μια επιστροφή στο μοντέλο εταιρικής σχέσης όταν αφορά τη διαχείριση των επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τον τομέα του investment banking. Αυτό ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι ηλεκτρονικά. Δύο ψήφοι λείπουν μία έκκληση ψηφοφορία. Εγκρίνεται 28 υπέρ 16 κατά. Εν τέλει εγκρίθηκε το σύνολο της συμβαστικής τροπολογίας M. Περνάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία N, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική O, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική P, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Q. Όχι, συγγνώμη. 437 πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα. Για την παράγραφο 25. Τροπολογία 437 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Q σε δύο τμήματα. Με συγχωρείτε λέει πρόεδρος. Πρωτότυπο κείμενο της παράγραφος 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Q πρωτοτμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ Ποιο είναι όμως το δεύτερο τμήμα. Συγγνώμη, δεν παρουσιάζεται πάρα πολύ καλά αυτή η συμβαστική τροπολογία στο κείμενο να σε εξηγήσω εδώ τι συμβαίνει. Έχουμε τη φράση να προβλέπετε όπου είναι αναγκαίο η δυνατότητα να υπάρχει μια νομική διαχώρηση όσον αφορά μια τράπεζα προκειμένου να αντιμετωπίσει χρεοκοπία, ενδεχόμενη χρεοκοπία. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει αυτή τη φράση, χωρίς, μάλλον το πρώτο τμήμα δεν έχει αυτή τη φράση, το δεύτερο την περιλαμβάνει. Περ, κατά, Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται όντως. 19 υπέρ και 26 κατά. Το τμήμα λοιπόν αυτό απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 447 υπέρ κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Όντως απορρίπτεται 20 υπέρ, 24 κατά. Περνάμε τώρα στην 448 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 449 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 450 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 451 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν σε ακούμε το μικρόφωνο παρακαλώ. Μετά 451 δεν πρέπει να ψηφίσουμε και το πρωτότυπο κείμενο το αρχικό. Ναι, αλλά ψηφίσαμε την 450, λέει ο Πρόεδρος. Η 451 απορρίφθηκε. Ακριβώς επειδή ψηφίσαμε 450, δεν έχουμε να ψηφίσουμε τώρα για το αρχικό κείμενο. 461 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 462 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 464 υπέρ κατά αποχές Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι κάνει το ΕΛΚΑ. Μπορούμε να ελέγξουμε για 464. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την 464. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ, 26 κατά. 463 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην 466 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 467 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία S υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 474 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 476 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 475 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Περνάμε στις 480 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 481 υπέρ, συγγνώμη. 481 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 483 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 484 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 485 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τα καταφέραμε. 486 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στις αιτιολογικές σκέψεις. Αιτιολογική σκέψη α. Έχουμε τέσσερις τροπολογίες εδώ. Βέρνερ, αφορά τις δικές σου τροπολογίες. Κύριε Λάγκεν, μ' ακούτε. Ελπίζω τουλάχιστον. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει ζητήσει να πούμε ότι είναι συμβατές οι τροπολογίες. Ναι, είναι περίπου συμβατές, είναι ήμι συμβατές. Ε, Νομίζω ότι η τροπολογία 9 του κυρίου Γκοζές διορθώνει τους αριθμούς. Μια στιγμή περίμενε, αλλάζει τους αριθμούς, αλλά αλλάζει, αφήνει τη διατύπωση όπως ήταν. Αν πρέπει να το ψηφίσουμε τώρα αυτό, το δεύτερο ήμιση της τροπολογίας του Βέρνε Λάγκεν και της ε, Βότμαν Κόρ, φαίνεται να είναι συμβατές στο περιεχόμενο, γιατί δεν έχουν σχέση με τα αριθμητικά στοιχεία. Αν απορρίψουμε την τροπολογία του κύριου Γκοζές, Αρλίν, ψηφίζουμε τις τροπολογίες, όχι αυτό που νομίζουμε ότι είναι αλήθεια. Συγγνώμη για να το ξεκαθαρίσω τεχνικά εδώ πέρα αν θεωρήσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει, ε, το έχει υπολογίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι γεγονός. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τους υπολογισμούς, ε, ε, είτε το υπερψηφίζεις είτε το καταψηφίζεις. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις άλλα στοιχεία από αυτά που υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τεχνικά δεν είναι συμβατή, βέβαια μπορείτε να το καταψηφίσετε άμα θέλετε. Ε, κάνε λίγο υπομονή ναι, αλλά δεν μπορείς να αλλάζεις τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν θες να το καταψηφίσεις, καταψηφίσέ το. Τι θα πεις ότι άλλα βρήκε η μελέτη της Επιτροπής. Πολιτικά δεν έχω πρόβλημα. Είναι τεχνικό το ζήτημα. Σου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω κάνει έναν υπολογισμό. Εσύ τον αφισβητείς. Να το καταψηφίσεις άμα θέλεις. Πού το βρήκατε αυτό το ποσό. Τεχνικά δεν ταιριάζει. Κάπως πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί τροπολογιών που λειτουργούν καλύτερα και νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει θέμα. Και επιστήσαμε την προσοχή σε αυτό. Είναι κόστος ή κρατική ενίσχυση που χορηγείται. Δηλαδή η κυρία Βόρτμαν Κόρ, ο κύριος Φέρμπερ, και ο κύριος Λάγκεν τι ε, λέγουν στις τροπολογίες τους. Και αν δεν θεωρείται κόστος αλλά κρατική ενίσχυση ε, και βάζετε όλα αυτά τα επιπλέον για το πώς δαπανήθηκαν. Η εναλλακτική λύση είναι να ακολουθήσουμε αυτό που λέει ο Ζαν Γκοζές και να αλλάξουμε το ποσόν ε, για το κόστος. Αυτό είναι το θέμα. Ε, κυρία Μακάρθη. Εντάξει, υπάρχουν κάποια ζητήματα, να τα ψηφίσουμε, να δούμε πώς θέλουμε να ψηφίσουμε και μετά το βλέπουμε στην Ολομέλεια. Αν είναι τεχνικές οι προσαρμογές, αν αυτό μας ε, προβληματίζει, το βρίσκουμε στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι έχουν καλό περιεχόμενο τροπολογίες, έχουν ουσία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν την ουσία. Ως Σαγετ, ένα μικρό θέμα μπορεί να επιδεινώσω την κατάσταση. Να ρωτήσω κάποιους που ανησυχούν για όλα αυτά. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην κρατική ενίσχυση και το κόστος για το φορολογούμενο. Όχι, για να ξέρω, απλώ ρωτάω. Um, I think, to be honest, I... Ε, λοιπόν, το θέμα είναι ποιο είναι το πραγματικό κόστος το, και όχι εγγύηση, που δεν είναι κατά ανάγκη κόστος πάντα. Για να είμαστε ακριβείς, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο εγγύηση. Εν πάση περιπτώσει, ας προσπαθήσουμε τώρα να ψηφίσουμε τροπολογία νέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος. Right, that is, that, that is 19 in fact. υπέρ 24 κατά απερίφθη. Λοιπόν, τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία του Βερνέρ Λάγκεν, ε, ψήφι υπέρ, στο σύνολο της κατά αποχές εγκρίνεται. Now I... Και τώρα νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε ε, ως προσθήκη το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας της Κορίν Βόρτμαν Κόλ που αφορά σε αυτά που ζητάει η Επιτροπή ε, αναδιάρθρωση τραπεζών που λαμβάνουν βοήθεια. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα, Μάρκους Φέρμπερ, έχουμε καλύψει τη δική σου τροπολογία, η οποία και καταπίπτει Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι ψηφίσαμε τα πάντα ε, στο αρχικό κείμενο, εκτός από το κόστος που έχει γίνει ενίσχυση. Η λέξη cost έχει γίνει grant. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο, γιατί έτσι θα ανατρεπόταν αυτό που ψηφίσαμε τώρα στις τροπολογίες. Λοιπόν, θα το ξαναδούμε στην Ολομέλεια, αν χρειαστεί. Τροπολογία 10, ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Κάνετε πολύ φασαρία, σταματάω. Right, we're now going to amendment Ερχόμαστε στην τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο της 13. Καλά. Ορίστε. Εγώ βλέπω και τον Ζαμπόλ και την Ελίζα με ψηλά τον αντίχειρα, οπότε συνήθως εγκρίνεται. 16 πέ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 πέ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα, που πάμε...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 I think this is, this is, this is... Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σκέτο χάλι όλο αυτό και δεν συμφωνώ ότι καταπίπτουν όλα αν εγκριθεί η τροπολογία Dorfman, διότι και πάλι έχει καλό περιεχόμενο, έχει ουσία και το υπόλοιπο των τροπολογιών. Οπότε, αν εγκριθεί η τροπολογία Dorfman, λέμε ε, ότι δημιουργούμε ένα στενές κανονιστικό πλαίσιο με ε, υπερβολικό και ανάληψη κινδύνου και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ε, την τροπολογία Λάγκεν για πολύ μεγάλους τραπεζικούς τομείς και το κεφάλαιο μετοχικό equity capital. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε τότε την υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 ήταν αυτή η κυρία Βόρτμαν Κόλ, μπορούμε να ψηφίσουμε και την 18 ως προσθήκη. Το γνωρίζω, λέει η Πρόεδρος. Α, μάλιστα, ευχαριστώ. Και τώρα είσαι σάντουιτς ανάμεσα στο Βένερ και την Κορίν, λέει ο κύριος Λάμερς. Και τη 19. 18 ως προσθήκη, λοιπόν. Με αντικίνητρα. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Έχω χάσει και χρόνο από τη συζήτηση σήμερα το πρωί ε, της συνεδρίασης για να το κοιτάξω αυτό. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην τροπολογία του Μάρκους και αυτό που μέχρι τώρα ψηφίσαμε στην τροπολογία του Βέρνερ, τι είναι. Ο Φέρμπερ θέλει να βγει η υπερβολική περιπλοκότητα του γενικού τραπεζικού τομέα. Το υπόλοιπο καλύπτεται. It changes those wordings around complexity, so I suggest we... Δεν ξέρω αν θέλουμε να το ψηφίσουμε. Για την υπερβολική περιπλοκότητα. Ψήφι υπέρ. Those against abstentions, right. So, uh, Marcus is... Λοιπόν, ε, η τροπολογία του Μάρκους δεν εγκρίθηκε, η υπερβολική περιπλοκότητα παραμένει και αφού το λύσαμε αυτό πάμε στην τροπολογία του Ζαν για το real estate. Όσοι θέλετε λοιπόν αναφορά στην κτήματα αγορά ψηφίστε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε στην τροπολογία 27. Ψηφίπε κατά αποχές εγκρίνεται. Όλες αυτές είναι τώρα συμβατές. 28 είπε Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Δεν απορρίπτεται. Τι κάνουμε λέει η κυρία Μακάρθη με την 28. Όταν είναι μόνο του το ΑΕΛΚ δεν κερδίζει ψηφοφορίες. Θα το καταλάβετε αυτό καμιά ώρα. Σας παρακαλώ. Την 28 ψηφίζουμε. Ψηφίζετε όλοι. Πέρασε. Close vote. And that is rejected. Απορρίπτεται. 21 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. 29. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. μισό λεπτό 44, πού το βρήκα αυτό, όχι, 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 τώρα υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να πιω λίγο νερό γιατί έχω πνιγεί και όλα votes closed. Ψηφίσατε όλοι. 23 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Τώρα τι ήταν αυτό που ψηφίζαμε. Το 44. 42 Ψηφίπε. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε. Everybody voted. That's carried. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται με 27 ψήφους προς 15, 43 υπέρ. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχο. Έλεγχος. Α, προστίθεται και κάποιες ψήφοι, θα έχει δίκιο. Ναι. Τα καταφέρατε. Ναι, αλλάζουν γνώμη οι ομάδες, λέει η κυρία Μακάρθη, η δικιά σου συγκεκριμένα. 47 in favor. 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, Τώρα ψηφίσαμε τη 47 και εγκρίθηκε μάλιστα. 48 ψήφι πέ. Κατά. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ τη 48 ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται 20 προς 25. Η τροπολογία 50 ψήφι πέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα θέλετε να, εγκρίνουμε, να ελέγξουμε την 58 παρακαλώ. εγκρινεται εγκρίνεται 26-17 62 είπε κατά αποχές απορρίπτεται 59 είπε κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε τώρα στην 69 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 70. Ψηφίσατε. Απορρίπτεται 21-23. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος για την 72 παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 20-23. Η 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω με την ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. 81 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. No, no, κ. Λάγκεν. Ε, ας το ελέγξουμε λοιπόν. Μήπως έχει αλλάξει συμπεριφορά κανείς στην ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 υπέρ και 23 κατά. Καταπίπτει λοιπόν κύριε Λάγκεν μου. Ή 87 υπέρ. Κατά. Είναι δύσκολο. Ε, τώρα θέλει έλεγχο η 87. υπερ κατα ειναι δυσκολο τωρα θελει ελεγχο η 87 απορριπτεται 21 υπέρ 22 κατά. Η 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα πάμε στην 91 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ για την 93. So if you voted, and that's carried, 27-17. Εγκρίθηκε 27-17. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θέλετε έλεγχο. Ε, να ελέγξουμε 94, δεν σηκώνετε χέρια. Ψήφισατε όλοι πέρα. Εγκρίθηκε. 95 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά έλεγχος για την 97 παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι, πέρας. Καταπίπτει. 20-20, ισοψηφία. Και τώρα πάμε στην 96, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90... 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν τρία. Υπέρ. Τι εκατόν τρία λέει η κυρία Μακάρθη. Ναι, υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για την 103 γιατί τα έχω χάσει λίγο το ΕΛΚ τι κάνει υπέρ είναι ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά 21 υπέρ 22 κατά 104 υπέρ Και εδώ χρειάζεται έλεγχο. 104 ψηφίζουν. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται 23-21. 99 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι. Έλεγχος λοιπόν για την 105 παρακαλώ. Εμένα μου φαίνονταν σαν να έχει εγκριθεί όμως. Εγκρίνεται 24-20 ορίστε. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Citations, αιτιολογικές αναφορές. Τι θέλετε έλεγχο για την 106, παρακαλώ. Μια στιγμή. Ελέγχουμε την 106, κυρία Σγκουλάρ. Ψήφισατε όλοι. 26, 17. Εγκρίνεται. Τις αιτιολογικές αναφορές μπορούμε παρακαλώ να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Unblock. Μέχρι τέλους, μέχρι τη 12. Υπέρ. Κατά αποχές. Ωραία εγκρίνονται και αυτές. Όλες. Θέλουμε λίγο χρόνο να καταλάβουμε τι ψηφίσαμε. Όχι. Ξέρουμε όλοι τι ψηφίσαμε. Μπράβο μας. Ε, γιατί υπήρξαν τόσα επίμαχα σημεία. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε ομελέτα, έχουμε στραπατσάδ. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Yes, me. Oh. I think I'll go. Uh, closed. Right, that's the... Ωραία, 36 υπέρ και 3 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται και 4 αποχές. coordinators meeting in here. Right. Okay, we have a coordinator. Εδώ, σε λίγα λεπτά.